Thank you, Mr. President. Can you hear me? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ακούτε? Χθες. Η Βασίλισσα έγινε η μακροβιότερη μονάρχη στον Ομένο Βασίλειο. Mm. Ελπίζω και η Βρετανία αλλά και οι Μαλτέζοι και οι Κύπροι συνάδελφοι αλλά και άλλοι συνάδελφοι βέβαια που δεν ανήκουν στην κοινοπολιτεία να εκφράσουμε την